Καλημέρα. Παρακαλώ, καθίστε. Βάλτε τις κάρτες σας στο μηχάνημα, τις κάρτες ψηφοφορίας στο μηχάνημα που προβλέπετε για αυτές. Όπως αποφασίσαμε χθες, η συζήτηση για τις ε, ενεργειακές υποδομές αναβάλλεται. Γι' αυτό σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουμε με το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση καονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό για τις ε, συνθήκες τις υγειονομικές που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ντεμπρούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ σήμερα το πρωί. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας. Ε, συζητήσαμε μέσα σε ένα επικοδομητικό πνεύμα για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μας απάντησε στις ερωτήσεις που θέσαμε. Πραγματικά μας έδωσαν απαντήσεις για τις εφαρμογές των παρεκκλήσεων και πώς θα λειτουργήσει το όλο σύστημα. Ε, οι σχέσεις μας ήταν αγαστές λοιπόν. Για τις τροπολογίες 4, 5, 4, 5 και 6. Θα ήθελα να πω στους βουλευτές ότι αυτές οι τροπολογίες ε, έρχονται σε έμεση αντίφαση με τις συστάσεις της δικής μου ε, έκθεσης. Την ακυρώνουν και επομένως ζητώ από όλους όχι μόνο τις καταψηφίσουν, αλλά εάν οι τροπολογίες 4, 5 και 6 περάσουν, τότε εγώ θα καταψηφίσω την έκθεση και θα ζητήσω και από τους υπόλοιπους να την καταψηφίσουν. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σας. Τώρα, ας περάσουμε στην ψηφοφορία αυτού του κειμένου. Πρώτη τροπολογία, Α, θέλετε το λόγο. Συγγνώμη, δεν σας είδα. κυρία Σουλιέ. Κυρία Αντωνέσκου. Ναι ή όχι. Όχι. Κυρία Σουλιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως συνεργαστήκαμε καλά με την κυρία Ντεμπρέν. Την ευχαριστώ. ευχαριστώ που μας άκουσε κιόλα και μας έλαβε υπόψη της. Αναφέρθηκε σε τρεις α, τροπολογίες του κυρίου Φράνκο. Αυτές οι τροπολογίες αφορούν μόνο τις προθεσμίες. Δηλαδή την παράταση που είχε ήδη δοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2010. Θέλουμε λοιπόν στην έκθεση να επιτρέψουμε μια δεύτερη παράταση. Στην πραγματικότητα θέλω μια εναρμόνιση, δηλαδή να μην έχουμε μεταβατικές, επιπρόσθετες μεταβατικές περιόδους. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω τις τροπολογίες Φράνκο και θα ήθελα και οι συνάδελφοι να τις υποστηρίξουν, που επί της ουσίας ζητάνε περισσότερη εναρμόνιση και απλούστευση για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων. Ευχαριστώ. Δεν θα το συζητούσαμε το θέμα. Να σας εξηγήσω ότι για τις χώρες που δεν έχουν α, μάλλον, ε, αν αυτό αφορά και τα άγρια είδη, νομίζω θα καταστρέψει την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Για αυτές τις χώρες που έχουν αυτές τις εξαιρέσεις θα πρέπει να τις συνεχίσουν. Γιατί αλλιώς ε, θα έχουμε αποφάσεις οι οποίες δεν θα σκοτώσουν αρρώστιες που θα σκοτώσουν τα ζώα σήμερα, αλλά αύριο, μεθαύριο. Πολύ ωραία. Να ψηφίσουμε τότε. Ναι, να ψηφίσουμε την πρώτη τροπολογία, άρθρο 1, σημείο 2. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Άρθρο 1, σημείο 3. Δεύτερη τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τέταρτη τροπολογία. Είναι μία από τις επίμαχες τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρθρο 1, σημείο 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έκτη τροπολογία, άρθρο 1, σημείο 7. Όχι, όχι, συγγνώμη. Τρίτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Υιοθετείτε. Τροπολογία 6. Άρθρο 1, σημείο 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πολύ ωραία. Τώρα θα ψηφίσουμε το συνολικό κείμενο και καταρχάς την ε, τροποποιηθήσα έκθεση υπέρ ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εντάξει, λειτουργούν τα μηχανήματά σας. Α, δεν έχετε την κάρτα σας. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Θα σας μετρήσουμε ούτως ή άλλως, κυρία μου. Ψήφισαν όλοι ηλεκτρονικά. Ούτε εσείς έχετε την κάρτα σας. Δεν μπορώ να ψηφίσω ηλεκτρονικά, αλλά ψηφίσω καταφατικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 33 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Όχι, Καμία αρνητική ψήφος, μία αποχή. Υιοθετείτε. Και τώρα θα ψηφίσουμε τον ίδιο τον κανονισμό. Υπέρ. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Σταματάει η ψηφοφορία. Πέρας μάλλον της ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Σας ευχαριστώ. Όσοι δεν είχαν την κάρτα τους να μας το πούνε. Μπορεί να σηκώσετε το χέρι όσοι δεν είχαν την κάρτα τους. Εντάξει. Ε, σας έχουμε λάβει υπόψη λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. και για την εξαιρετική ποιότητα της έκθεσής της. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. που αφορά το ΣΥΤΕΣ. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση για την ε, συνεδρίαση την, της 15ης διάσκεψης των μερών του ΣΥΤΕΣ που θα γίνει στην Τόχα το Μάρτιο και που θα αποφασίσει διάφορα, διάφορες προτάσεις ε, ψηφίσματος. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο παρατήματα στο ΣΥΤΕΣ, το παράρτημα 1 όπου απαγορεύεται 100% το εμπόριο και το παράρτημα 2 όπου το εμπόριο ελέγχεται. Θα κάνουμε μια συζήτηση τώρα για διάφορα είδη, τον ερυθρό τόνο, την, τον ελεφαντά της Αφρικής, ε, την Πολική Αρκούδα, τον ε, Καρχαρία και το Σκυλόψαρο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ο κύριος Λάγκεντορφ είναι εδώ. Και τα μεγάλα λουροειδή, συγγνώμη, επίση. Ε, θα ξεκινήσουμε την κυρία Γιούζο, η οποία ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν ε, είμαι καθόλου εμπειρογνώμονας ε, για θέματα λίας, αλλά κυρία Φράγκα, που είναι συντονίστρια για θέματα λίας, μου ζήτησε να σας διαβάσω το κάτω σημείωμα για αυτό το ψήφισμα. Το πρώτο σημείο αφορά τον ερυθρό τόνο. Το εκτιμώντα 1 και η παράγραφο 4 της πρότασης ψηφίσματος μιλάει για αυτό το θέμα. Η... Η Επιτροπή για τα Τονοειδή του Ατλαντικού, ε, ΙΚΤΑ, στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου του 2009 α, θεωρεί ότι η βιομάζα γόνου του τόνου είναι κατώτερη από το 15% από ό,τι ήταν ε, στην ε, έναξη της περίοδου, στην του ψαρέματος ε, του τόνου. Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να μπει ο ρυθρός τόνος στο πρώτο παράρτημα του ΣΥΤΕΣ. Συμφωνήθηκε λοιπόν ότι ο ρυθρός τόνος πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ΣΥΤΕΣ για τη συμπερίληψή του στο παράρτημα 1. Και το σημείο 4 θα την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τον ερυθρό τόνο στο παράδειγμα 1 του ΣΥΤΕΣ, σύμφωνα με τους ε, στόχους της πρότασης. Αυτό είναι λάθος. Αυτό, αυτό είναι μια ερμηνεία από μη κυβερνητικές οργανώσεις και διορθώθηκε στην ιστοσελίδα. Επομένως, η έκθεση της ε, συνεδρίασης λέει ότι Δύο από τα κριτήρια δεν πληρούνται. Και σε ό,τι αφορά το τρίτο κριτήριο, όλα εξαρτώνται από τα λιεύματα που επιτρέπεται να ληφθούν. Η ετήσια συνάντηση του ΙΚΑΤ της Διεθνούς ε, Επιτροπής Διατήρησης για τον τόνο του Ατλαντικού λέει ότι μάλλον ε, αποφασίστηκε στη Βραζιλία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι συμβαλόμενο μέρος ότι Τα συνολικά αλλιεύματα τόνου θα είναι 350.000 τόνοι, ε, μείωση κατά 40%. Επίσης αποφασίστηκε για το 2011 να κάνουμε περαιτέρω μείωση 50%. Ε, επίσης, για τις, τα αλλιευτικά σκάφη, η περίοδος ψαρέματος θα μειωθεί κατά ένα μήνα. Η Επιτροπή ΙΚΑΤ συμφώνησε για ένα τάκ ε, του χρόνου που θα είναι κάτω από τους 15.000 τόνους. Γιατί η σύσταση που υιοθετήθηκε για 13.000 τόνους ε, ουσιαστικά συνάδει με, τις με τα επιστημονικά πορίσματα. Επομένως, θα πρέπει να ε, διαγράψουμε την παράγραφο 4. Σε ό,τι αφορά τους καρχαρίες, στο σημείο J, λέει, σε ό,τι αφορά τα, τους καρχαρίες και τα σκυλόψαρα, που είναι πάρα πολύ ευπαθή ήδη, λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών τους και της μεγάλης αλίευσης, ε, λόγω του ότι έχουν ε, βραδύ ανάπτυξη, αργοπορημένη οριμότητα, χαμηλή αναπαραγωγική ικανότητα κτλ. Και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα, τους καρχαρίες και τα σκυλόψαρα στο παράδειγμα 2. Αυτό το υπέβαλαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Σουηδία. Σημείο 6. Ε, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν ε, την καταχώρηση των πέντε ειδών καρχαριών ε, Σμύρνα Λέβινη, Σμύρνα Μοκάραν, Σμύρνα Ζαγκένα, Καρχαρίνους Πλομπέους και Καρχαρίνους Οψκούρους στο παράτημα 2 του ΣΥΤΕΣ με βάση την πρόταση του, των ΗΠΑ. Σημείο 7. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν την καταχώρηση του ωκεάνου χαρακτήρα καρχαρίνου Λογκυμάνου στο παράτημα 2 του ΣΥΤΕΣ σύμφωνα με την πρόταση των ΗΠΑ της Αμερικής. Θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή ότι είναι περίεργο που ο μόνο καρχαρία του οποίου η αλίευση απαγορεύθηκε από την ΙΚΑΤ είναι ο αλόπιος σας Και αυτό θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την πρόταση ή σε καμία άλλη πρόταση. Ε, είναι ένας καρχαρίας που πραγματικά είναι απειλούμενο είδος. Η λάμια επίσης δεν έχει ρυθμιστεί στο εσωτερικό του ΣΥΤΕΣ. Επίσης αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να αναμένει την τελική απόφαση για όλα τα είδη που αλλιεύουν τα ληφτικά σκάφη. Θα πρέπει να περιμένουμε ε, να λάβουμε μια επιστημονική έκθεση, η οποία ετοιμάζεται από τους εμπειρογνώμονες, ούτως ή άλλως ε, ετοιμάζεται κάθε χρόνο, για το αν θα συμπεριληφθούν κάποια είδη στα παρατήματα ή όχι. Αυτό θα αποφασιστεί στις 7 με 10 Δεκεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Ε, θα έχουμε έτοιμη αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να σας πω ευχαριστώ και εκ μέρους των συντονιστών. Ευχαριστούμε κύριε Γιούζο. Δίνω το λόγο στον Κρίστε Δης. Συμφωνώ με αυτά τα οποία ο κύριος Ντέιβις. Ε, συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Προτείνονται οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη ΣΥΤΕΣ. Γνωρίζω ότι οι βουλευτέ εμεί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε πολύ μικρή επιρροή σε αυτά τα οποία γίνονται και τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται ε, μεμονωμένα, παρότι υπάρχει συντονισμό μεταξύ του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω δεν έχει επίσημη συλλογική παρουσία στην ΣΥΤΕΣ. Θα ήθελα να ακούσω όμω και κάποια σχόλια εκ μέρου τη επιτροπή ή των εκπροσώπων του Συμβουλίου σχετικά με του στρατηγικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε μαζί τους να συζητήσουμε τις προτεραιότητες και να τους ζητήσουμε να σκεφτούν τα σημεία που μας ανησυχούν. Αν υπάρχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, θα μπορούσε να κάνει κάποια παρέμβαση τώρα ή και αργότερα στη συζήτησή μας, γιατί θα μας βοηθούσε αυτό. Ευχαριστούμε, Κρίς, λέει η Πρόεδρος, αλλά δεν ήταν εκπρόσωπος της Επιτροπής εδώ όταν προλίγου τον αναζητήσαμε για να λάβει, το, να λάβει μέρος στη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ακόμη εξάλλου εκπρόσωπος της Επιτροπής, άρα δεν μπορώ να ικανοποιήσω το έτοιμά σας, πράγμα το οποίο με λυπεί. Να δώσω λόγο στον κύριο Σερμπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω το ψήφισμα αυτό και ελπίζω να μπορέσουμε να το εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, έχω ένα ερώτημα. Αρχικά, είχε αναφερθεί 22 Δεκεμβρίου ως ημερομηνία που θα το συζητούσε το Συμβούλιο. Αλλά νομίζω ότι έχει βγει από την ημερήσια διάταξη δεν θα το συζητήσει λοιπόν η Σουηδική Προεδρία και θα μεταφερθεί στην Ισπανική Προεδρία. Επίσης, θα ήθελα να αναρωτήσω τη γραμματεία της Επιτροπής μας αν μπορεί να διασφαλίσει ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια με βάση τις προφορικές ερωτήσεις και την ε, έγκριση του ψηφίσματο. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει πριν γίνει η συζήτηση στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, γιατί θα ήταν κρίμα να καθυστερήσουμε εμείς και να φτάσει η δική μας απόφαση μετά το Συμβούλιο. Επίσης θα ήθελα να προσέξουμε ιδιαίτερα τον βόρειο ερυθρό τόνο. Χαίρομαι που αναφέρεται εδώ αυτό το είδος. Και ένα πρόβλημα έχουμε με το Συμβούλιο, διότι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πείσαμε το Σεπτέμβριο ότι ο ερυθρός τόνος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της ΣΥΤΕΣ αλλά η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου ψήφισε κατά αυτή τη πρόταση, παρότι ο πρόεδρο Σαρκοζή πιστεύει ότι πρέπει να σταματήσει η ελίευση του ερυθρού τόνου. Ο Γάλλο εκπρόσωπο ε, στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου ψήφισε κατά τη συμπερίληψη του ερυθρού τόνου στο παράρτημα 1 τη ΣΥΤΕΣ. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους, ιδιαίτερα από τις μεσογειακές χώρες, όχι μόνο να υπερψηφίσουν αυτό το ψήφισμα, αλλά και να κάνουν ό,τι μπορούν και να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τους συναδέλφους τους στα εθνικά κοινοβούλια, για να διασφαλίσουμε ότι ο ερυθρός τόνος δεν θα γίνει το είδος το οποίο θα εκλείψει λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Εκτός από τις ποσοστώσεις που είναι πολύ υψηλέ, πρέπει να πούμε ότι είναι και πολύ υψηλό το ποσοστό της παράνομης αλίας και θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιο έλεγχο επί των εμπορικών συναλλαγών και αυτό μπορεί να γίνει ε, μόνο μέσω του παρατήματος 1 της ΙΤΕΣ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κερμπραντή, θα ήθελα ένα σχόλιο απλώς να κάνω εν είδη διευκρίνηση. Η ψηφοφορία όντω προβλέπεται στην Επιτροπή περιβάλλοντο τέλη Ιανουαρίου 2010 και προβλέπεται για την Ολομέλεια η ψηφοφορία το Φεβρουάριο. τροπολογίε πρέπει να κατατεθούν μέσα στο Δεκέμβριο. Άρα όντω έχουμε μια καθυστέρηση. Ο κ. Σλούτερ. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να υποστηρίξω το ψήφισμα αυτό. Πιστεύω ότι γενικά είναι καλό το ψήφισμα και εγώ συμφωνώ ο ερυθρός τόνος να συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα 1 διότι είναι είδος ε, που βρίσκεται σε κίνδυνο ε, και είναι τόσο κακή η κατάσταση αυτού του είδους ε, που πρέπει οπωσδήποτε να απαγορεύσουμε το εμπόριο τώρα αν δεν το κάνουμε τώρα, δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το είδος ερυθρός τόνος, ε, τόνους, θύνους. Επίσης, ε, θα ήθελα να αναφέρω για τον Καρχαρία, συγκεκριμένα για τον Καρχαρίνους πλουμπέους, που επίσης ε, αναφέρεται στο κείμενο ότι οι μέθοδοι αλληλείας που χρησιμοποιούνται δεν είναι αποδεκτές. Σε ορισμένες ασιατικές χώρες θεωρούν ότι τα πτερήγια του έχουν μαγικές δυνάμεις και μπορούν ε, να επιδράσουν πολύ θετικά στον οργανισμό και κόβουν τα πτερήγια του καρχαρία και τελικά αφήνουν τον καρχαρία να πεθάνει στο νερό με κομμένα τα πτερήγια. Ακόμη και αν δεν βρίσκεται λοιπόν σε άμεσο κίνδυνο θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε σε αυτό το παράδειγμα. Κάτι άλλο που νομίζω ότι λείπει σε αυτή την έκθεση είναι ο Ευρωπαϊκός Λίγκας, ο Links Links. Όπως επίσης και ο Λίγκας της Ιβηρικής και ο Bobcat, ο Αμερικανικός Λίγκας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να αφαιρέσουν αυτό, αυτά τα από τον ε, κατάλογο της ΣΥΤΕΣ θεωρούν ότι δεν είναι είδο ε, που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αλλά δεν μπορεί να διαφοροποιήσει κανεί τον Αμερικανικό link από τον Ευρωπαϊκό link, Άρα ο link ο Αμερικανικό δεν μπορεί να ε, αφαιρεθεί από τον κατάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα αφαιρεθεί ο Αμερικανικό link από τον κατάλογο, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εμπόριο και ευρωπαϊκού Λίγκα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο. Οι Αμερικανοί κάνουν ε, μια προσπάθεια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ειδών, αλλά μέχρι ότου καταφέρουν να κάνουν τη διαφοροποίηση, Εμεί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καταψηφίσουμε αυτή την πρόταση των Αμερικανών. Σα Σας ευχαριστώ. Και έχουμε τώρα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοντά μας. Τον καλωσορίζουμε. Συγγνώμη που με το που μπαίνετε μέσα σας ε, πιάνουμε από το λαιμό, αλλά αρκετοί συνάδελφοι σας περίμεναν για να ακούσουμε τη στρατηγική της Επιτροπής. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τη στρατηγική της Επιτροπής. Καλή σας μέρα. Γνωρίζετε ότι οι προετοιμασίες για την COP15 από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγονται σε δύο στάδια. Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2009 Υπευλήθησαν προτάσεις, ε, αυτές οι προτάσεις λέει τις οποίες θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην COP15. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις, έχουν προταθεί και από άλλα μέρη και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο καθορισμού της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις προτάσεις που υπευλήθησαν από άλλα μέρη. Αυτή είναι μια κλασική διαδικασία στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 302, το πρώην άρθρο 302 και η Επιτροπή προετοιμάζει τώρα την πρότασή της προς το Συμβούλιο. Αυτή η πρόταση θα εξετάσει όλες τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τα άλλα μέρη και θα λάβουμε θέση είτε για όλες είτε για τις πιο σημαντικές από τις προτάσεις αυτές. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα θέματα που είναι πολιτικά ευαίσθητα όπως είναι η πολική άρκτος, ο ερυθρός τόνος, οι ελέφαντες, το εμπόριο ελεφαντοστού κλπ. Σε αυτό το στάδιο κάνουμε ακόμη συζητήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις μας. Άρα δεν μπορώ να σας πω και πολλά πράγματα προς το παρόν. Το ψήφισμά σας φτάνει λοιπόν σε μια ιδιαίτερα κατάλληλη χρονική στιγμή, γιατί θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μέτρο του δυνατού για τα διάφορα θέματα τα οποία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόλις έχει διαμορφωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ελπίζουμε, ή αρχές Ιανουαρίου, θα αρχίσουμε και επισήμως τις συζητήσεις στο Συμβούλιο υπό Ισπανική Προεδρία. Και θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να είναι έτοιμη για την ΚΟΠ το Μάρτιο του 2010. Ακόμη λοιπόν διεξάγονται συζητήσει στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαμορφωθεί η πρόταση τη Επιτροπής για τα βασικά θέματα. Και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολες αυτές οι συζητήσεις. Συμπεριλαμβάνουν τον ερυθρό τόνο, τούνους, την πολική άρκτο, τους ελέφαντες κλπ. Δυστυχώς αυτά έχω προς το παρόν να σας πω για το στάδιο της προετοιμασίας. Δεν έχουμε ακόμη καθορισμένη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα πρέπει να περιμένουμε και για τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Chris Davis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής να μας πει ε, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ΣΥΤΕΣ, δηλαδή πώς θα εξασφαλίσετε μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΣΥΤΕΣ και τι θα γίνει αν δεν έχουμε μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω ακούσει το, στο παρελθόν ότι αν δεν μπορούμε τελικά να έχουμε συμφωνία θα απόσχουμε. Μπορείτε να μας πείτε σε μια διάσκεψη όπως τη ΣΥΤΕΣ πώς υποβάλλεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε μια νομική προσωπικότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας ρωτώ πώς υποβάλλεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα θέματα αυτά τα οποία έχουμε στο ψήφισμα το δικό μας, ε, θέλω να πω ότι έχουν σχέση με τα πολιτικά θέματα που αφορούν τον ερυθρό τόνο. Όλοι γνωρίζουμε τα τα θέματα αυτά και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, ότι υπάρχει ε, ε μια μειοψηφία που προς το παρόν δεν επιτρέπει την ψήφιση ε, αυτού του θέματος στο Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι και η Ισπανία και άλλες χώρες διαφωνούν. Και ε, εκτός από αυτό το θέμα για τον ερυθρό τόνο και το θέμα του εμπορίου ελεφαντοστού είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι πολιτικά ευαίσθητο. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχετικά με τη διαδικασία και το ποια θέση ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΣΥΤΕΣ, όντως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι μέλος της ΣΥΤΕΣ. Οι ΣΥΤΕΣ είναι μία από τις παλαιότερες συμβάσεις όπου δεν μπορούσαν ε, να γίνονται μέρη περιφερειακές ε, οργανώσεις κρατών και έχουμε καθεστώς παρατηρητού ως κοινότητα. Βεβαίως αυτό δεν μας έχει αποτρέψει να μιλάμε με μία ενιαία φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι δηλαδή δεν είναι μέλος της ΣΥΤΕΣ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προεδρία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπώντας τα συμφέροντα της ε, κοινότητας και των κρατών μελών. Η διαδικασία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση στο Συμβούλιο όπου διατυπώνεται αυτό το οποίο η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να είναι η θέση της κοινότητας και το Συμβούλιο εγκρίνει αυτή τη θέση και το Συμβούλιο ηγείται των διαπραγματεύσεων. Η Προεδρία ηγείται των διαπραγματεύσεων στην ΣΥΤΕΣ. και στη συνέχεια εν γέννη η Προεδρία είναι αυτή που εκφράζεται εκ μέρους των κρατών μελών. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν επιλύονται στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου και ορισμένα από αυτά πρέπει επιτόπου να επιληθούν. Θα φροντίσουμε όμως για τα σημαντικά θέματα να υπάρχει με τον α ή β τρόπο κοινοτική θέση. Σε ορισμένα σημεία μπορεί να επιλέξουμε και την αποχή. Δεν έχω ακόμη σαφή εικόνα. Είναι κάτι όμως που μπορεί να συμβεί. Πρέπει πρώτα να δούμε όμως τι θα γίνει στο Συμβούλιο. και αν υπάρχει στο Συμβούλιο κάποια θέση, αν δεν υπάρχει πλειοψηφία ή αν υπάρχει κάποια ελέγχουσα μειοψηφία, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ ακόμη να σας ε, προβλέψω το αποτέλεσμα των συζητήσεων. Προς το παρόν, απλώς εξετάζουμε αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε για να καταλήξουμε σε κάποια θέση ε, της κοινότητας. Αυτό κάνουμε συνήθως όχι μόνο για τις ΣΥΤΕΣ, αλλά γενικά για τη θέση της ε, κοινότητας ε, σε διεθνείς περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις τέτοιου είδους. Επανέρχομαι τώρα σε αυτά τα οποία και εσείς αναφέρετε ως πολιτικά ευαίσθητα θέματα και το θέμα του ερυθρού τόνου. Ξεκινάμε από ένα έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά την Επιτροπή, τη Διαχειριστική Επιτροπή ε, ΣΥΤΕΣ της 21 Σεπτεμβρίου ακόμη επιφυλασσόμεθα για το αν ε, θα υποστηρίξουμε την πρόταση να συμπεριληφθεί στο παράρτημα 1. περιμέναμε την 21η συνάντηση της ECALT, της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τονοειδών, πριν από δύο εβδομάδες και περιμένουμε να εξετάσουμε και περαιτέρω επιστημονικές πληροφορίες που ενδεχομένως ε, θα τεθούν στη διάθεσή μας ε, σε αυτό το διάστημα, ήδη δηλαδή από το Σεπτέμβριο που πέρασε μέχρι τώρα. Ξέρουμε τα αποτελέσματα στο Ρεσίφε. Η ερμηνεία που μπορεί να δοθεί ποικίλει. Μπορεί να πει κανείς ότι ελήφθησαν κάποια θετικά μέτρα. Η ICAT, Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Ειδών του Ατλαντικού, έλαβε θετικά μέτρα για τη διατήρηση των ειδών. Είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα θετικό βήμα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε πριν. Παράλληλα, αρκετές σημαντικές αποφάσεις έχουν αναβληθεί για την επόμενη χρονιά, για, την, ε, για τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα, παραδείγματος χάρη. Και η Επιστημονική Επιτροπή της ICAT έλαβε εντολή από την ICAT να κάνει μια ανάλυση σχετικά με τα κριτήρια της ΣΥΤΕΣ, για το αν πληρούνται δηλαδή οι προδιαγραφές για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο του παραδείγματος 1 της ΣΥΤΕΣ. Έγιναν πολλές τέτοιες συζητήσεις γύρω στον Αύγουστο-Σεπτέμβριο και το θέμα είναι το αν τα κριτήρια συμπερίληψης στο παράρτημα 1 πληρούνται. Πάντοτε γίνεται μια τέτοια εξέταση για να επιβεβαιώσουμε το αν κάποιο είδος πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο 1, στο παράρτημα 1, στο παράρτημα 2. Η Επιστημονική Επιτροπή της ΆΕΚΑΤ ε, Έδωσε την γνωμοδότησή της τον Οκτώβριο και το εξετάζουμε τώρα και το λαμβάνουμε υπόψη μας για να αποφασίσουμε το αν θα υποστηρίξουμε την πρόταση του Μονακό ή όχι. Το συζητούμε και στις υπηρεσίες της Επιτροπής και αυτή τη στιγμή που το συζητάμε εμείς εδώ είναι ακριβώς αντικείμενο διαπραγμάτευση σε πολλά βήματα. Δεν μπορώ λοιπόν να προβλέψω το τι θα προκύψει από τις συζητήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα είδη που αναφέρθηκαν, για την πολική άρκτο παραδείγματο χάρη. Γίνεται παράλληλα με την τωρινή συνεδρίαση σήμερα στο κτίριο Μπορσέτ μια συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής για το θέμα της πολική άρκτου θα συζητηθεί το θέμα της πολιτικής άρκτου, παρουσία του εκπροσώπου του Καναδά και της Γρινλανδίας και θα γίνει και βίντεο διάσκεψη με κάποιον στις Ηνωμένε Πολιτείε ταυτόχρονα για να ακούσουμε τα υπέρ και τα κατά της πρότασης των Ηνωμένων Πολιτειών για να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν είναι λοιπόν τελική η θέση της Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για τους ελέφαντες και το ελεφαντοστούν. Στην COP14 πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι συμμετέχει και πάλι τα ίδια θέματα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και τελικά βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση Και ακούγονται στις προτάσεις που υπευλήθησαν και από τις δύο πλευρές, Ζάμπια και Τανζανία αφενός και συνασπισμός άλλων χωρών αφετέρου, Κένιας κλπ. Ακούσαμε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Και είναι ακόμη πρόωρο το να κάνουμε προβλέψεις για το ποια θα είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη. Είναι ένα θέμα που ίσως πρέπει σε κάποιο βαθμό να το αφήσουμε ανοιχτό για να υπάρχει περιθώριο ελιγμών για να γίνει συζήτηση μεταξύ των μερών στην COP15 για να δούμε πώς μπορούν να συμφιλειωθούν οι διεστάμενες απόψεις στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ την Κομισιόν για τις εξηγήσεις, λέει ο κ. Θέλω πραγματικά να συζητήσουμε με την Ισπανική Προεδρία το θέμα του ερυθρού τόνου, αλλά δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η συζήτηση αν η απόφαση του Συμβουλίου έχει ήδη ληφθεί τη στιγμή που θα το συζητήσουμε στο Ολομέλεια. Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα της Προεδρίας, πότε θα αποφασίσει το Συμβούλιο ε, για τα θέματα του ΣΥΤΕΣ επίσημα και πότε οι συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου θα λάβουν χώρα. <clears throat> Γιατί δεν θα ήθελα οι εμπειρογνώμες του Συμβουλίου να αποφασίσουν πριν εμείς συζητήσουμε το θέμα αυτό με το Συμβούλιο. Μια άλλη τεχνική ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, ότι χρειάζεται περίπου έξι μήνες μετά την απόφαση της Ντόχα. Έξι μήνες για να αποφασιστούν τα πάντα. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε για τις ΣΥΤΕΣ να βάλουμε τον ερυθρό τόνο στο παράρτημα 1, θα χρειαστούν άλλοι 6 μήνες. Δηλαδή, θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Δηλαδή, 10 περίπου μήνες, ας πούμε, της αλληλευτικής περίοδου του 2010 θα έχουν περάσει πριν γίνει κάτι για τον ερυθρό τόνο. μια παρατήρηση για το σχόλιο του εκπροσώπου της Επιτροπής για τις πολιτικές αρκούδες. Διαρωτώ με, μπορείτε να μας δώσετε κάποια ένδειξη της αξιολόγησης επιστημονικών στοιχείων για τον αριθμό των πολιτικών αρκούδων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιοι που έχουν επιφυλάξει, έχουν λένε ότι υπάρχει μείωση του αριθμού. Και αυτό Άλλοι ε, λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με ανθρώπους. Τι συμβαίνει ακριβώς. Monsieur le représentant de la Commission, si vous voulez bien répondre. Commission, θα ήθελα να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Ευχαριστώ. President, um, on the, the, the... Για τη χρονική στιγμή για τις συζητήσεις στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Όπως θυμάμαι εγώ τα πράγματα, η Ισπανική Προεδρία θα ήθελε να έχει μια πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και μια δεύτερη συνάντηση κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Τώρα φυσικά νόημα έχει μόνο τότε να έχουμε μια συνάντηση ομάδας εργασίας του Συμβουλίου όταν θα υπάρχει πρόταση της Επιτροπής Επιτραπέζης. Ο σχεδιασμός μας είναι να εκδοθεί το δυνατόν, να υποβληθεί το δυνατόν νωρίτερα, ελπίζοντας κατά τα τέλη αυτού του έτους. Αν όχι, πολύ νωρίς ε, κατά τις αρχές Ιανουαρίου 2010 να υποβληθεί η πρότασή μας. Για το ακριβές χρονοδιάγραμμα είναι πολύ δύσκολο να πω οτιδήποτε και να σας ενημερώσω σε αυτή τη φάση. Είναι όμως σαφές ότι θα υπάρξει ένας αριθμός συναντήσεων στο, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και σε σχέση με την απόφαση επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ληφθεί πριν από τη συνάντηση του ματιού 2010 της ΚΟΠ. Τώρα έχουν υπάρξει άτυπες φυσικά συζητήσεις με εκείνα τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται ήδη για να αποκομίσουμε εντύπωση ποια είναι η στάση τους ή η τοποθέτησή τους επ' αυτών. Συναντήσεις με ΜΚΟ για να υποβληθούν οι απόψεις τους για διάφορα θέματα. Αρκετές άτυπες συνεδριάσεις έχουν γίνει σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα το ερώτημα πότε θα ήταν δυνατόν να, έχουμε, να αρχίσει να ισχύει το παράτημα ένα όσον αφορά την απόφαση. Από ό,τι θυμάμαι για την για ημερομηνία θα πρέπει να το ξαναδώ το θέμα αυτό όμως. Μία περίοδο 18 μηνών να έχει προταθεί πριν από την έναξη σε ισχύ. Αλλά όπως είπα πρέπει να το επανελέγξω αυτό. Δεν θα άρχιζε να ισχύει άμεσα. Με άλλα λόγια. Θα επανέλθω όμως για να σας ενημερώσω γι' αυτό όταν θα το έχω ελέγξει. Ένας, μια πρόταση που θα συνοδεύεται και από μια πρόταση ψηφίσματος. Τώρα για τις πολιτικές αρκούδες, ρωτήσατε ποιος είναι ο αριθμός τους. Δυστυχώς ε, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να έρθω σε επαφή και να διαβιβάσω την ερώτησή σας σε παίοντες. Ευχαρίστως όμως από πλευρά τους θα σας διατεθούν τα στοιχεία. Ένα από τα θέματα που συζητείτε είναι σε ποιο εύρος το εμπόριο δημιουργεί προβλήματα για τις πολικές αρκούδες. Και είναι ένα από τα σημαντικά φυσικά κριτήρια να αποφασίσουμε για το αν σε αυτή την περίπτωση θα αναβαθμίσουμε από το παράτημα 1 στο παράτημα 2 τις ε, πολικές αρκούδες. Είναι το εμπόριο, εκείνο το πρόβλημα που δημιουργεί προσκόμματα θα ε, δικαιολογεί το μία αναβάθμιση λόγω αυτού από το παράτημα 1 στο παράτημα 2 των πολικών αρκούδων. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε από τα κράτη-μέλη. Να εξεταστεί αυτό προσεκτικά. Να δούμε λοιπόν αν απειλούνται οι πολικές αρκούδες λόγω εμπορίου, λόγω των ε, εμπορικών ε, ε, εξελίξεων ή κυρίως λόγω αυτών θα το δούμε αυτό και φυσικά είναι ένα στοιχείο το οποίο εξετάζουμε μέσα στο πλαίσιο της κανονικής ανάλυσης που πρέπει να γίνεται όταν αποφασίζουμε την εγγραφή, την καταχώρηση και με βάση τις συγκεκριμένες προτάσεις. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το στοιχείο του εμπορίου στην μείωση του αριθμού αυτών των ειδών. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Υπενθυμίζω τις τροπολογίες. Θα πρέπει να τις καταθέσετε πριν τις 8 Δεκεμβρίου. Θα ψηφίσουμε θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΜΒΗ με ένα ερωτηματικό στο τέλος Ιανουαρίου και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια πάλι ερωτηματικό το Φεβρουάριο του 2010. Πάω στο επόμενο σημείο της σημερισίας διάταξης, ε, που είναι ένα προφορικό ερώτημα, το οποίο θα θέλαμε να υποβάλουμε προς το Συμβούλιο για την στρατηγική και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσκεψη των μερών. Έχετε στο φάκελό σας το σχέδιο ερώτησης, που είναι πάρα πολύ μετρημένη ερώτηση και πάρα πολύ ισορροπημένη. Θα ήθελε κανένας να πάρει το λόγο για αυτό το σχέδιο ερώτησης. No. Oui. Personne ne veut la parole. Κανείς το λόγο. Είναι πολύ εύκολο να το διαβάσει κανείς. Τρεις γραμμές είναι για όσους δεν το διαβάσατε το λέω. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό το ερώτημα. Μια και το εμβαθύναμε τόσο πολύ. Ποιο είναι υπέρ, Ποιο είναι κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Θα θέσουμε αυτό το ερώτημα από τη μορφή που το λάβαμε. Πάμε στο επόμενο σημείο τώρα. Που αφορά τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Είναι ένα σχέδιο τροποποίησης της οδηγίας 2001 93 εκα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ματίας. Την κυρία Ματίας. <laughs> Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μια ευκαιρία αυτή, εξαιρετική ευκαιρία ε, για να ανταλλάξουμε τις πρώτες απόψεις για αυτή την πρόταση οδηγίας. Αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι μια πρόταση οδηγίας προς το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έναρξη σε ισχύ όσον αφορά τα ψευδεπίγραφα φάρμακα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα τομέα όπου μας χρειάζονται ακόμα στοιχεία αξιόπιστα, αυστηρά αξιόπιστα στοιχεία για να ξέρουμε ποιο είναι το εύρος αυτού του φαινομένου. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να κάνω, να σχεδιάσω ένα γενικότερο πλαίσιο, κυρίω για να ακούσω και τις προτάσεις και τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων, αλλά να κάνω όμως να παρουσιάσω ένα πλαίσιο για τις δικές μου προτάσεις για αυτό το θέμα. Έχουμε λοιπόν εδώ από πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θεωρούν ότι ένα ποσοστό των φαρμάκων αυτών είναι ψευδεπίγραφα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μικρό ποσοστό όταν συγκρίνεται με το ποσοστό που χρησιμοποιείται παγκόσμια. Όμως αυτό το οποίο εδώ καταφέραμε να κάνουμε θα είναι σημαντικό και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο μέλλον για άλλες περιοχές όπου είναι μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό, αλλά κυρίως για να υπάρξει η ασφάλεια, η εγγύηση από πλευράς της κυκλοφορίας αυτών των φαρμάκων. Αυτά τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή για την διανομή, δηλαδή την πώληση στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, κάνουμε λόγο και για μεγάλα στοιχεία. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτή η πρόταση να ληφθεί υπόψη για τη διαχείριση και αντιμετώπιση της ίδιας της υγείας των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουν συγκίτρια για αυτό το σχέδιο όταν είχε υποβληθεί στην Ευρωβουλή και πρέπει να πω ότι άκουσα πάμπολους εμπλεκόμενους σε αυτή την ε, ακρόαση και διαδικασία σε όλη την αλυσίδα διανομής και εμπορίας ακούσαμε και τις εκθέσεις και τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών. Και αυτό είναι ένας διάλογος όπου έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα και γι' αυτό συζητούμε αυτό το θέμα και ανταλλάσσουμε απόψεις και θέλω σήμερα να ακούσω τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα σε σχέση με τα θέματα που έχουμε μπροστά μας. Κάποια θέλω να υπογραμμίσω μόνο γιατί δεν μπορώ όλα να τα καλύψω. Να υπογραμμίσω κάποια που θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπήρχαν θέσεις που διαμορφώθηκαν για αυτές τις ε, υποθέσεις, για αυτά τα ζητήματα. Αυτή η οδηγία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, πιστεύω εγώ, έναν ορισμό του τι είναι ψευδεπίγραφο προϊόν, προϊόν μαϊμού, για να μην ε, νομοθετούμε εν κενό να μην δημιουργούμε δηλαδή νομοθεσία για κάτι που δεν έχουμε καθορίσει καλά. Επίσης, ορισμοί του ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εμπλέκονται στις ε, διαδικασίες αυτές. Από την άλλη πλευρά, η ασφάλεια των, η υγεία των ασθενών είναι προτεραιότητα και γι' αυτό πρέπει να έχουμε διπλή νομική βάση και να μην μείνουμε, ας το πω έτσι, μόνο στο άρθρο 95 όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά και τη λειτουργία της, αλλά και το 152 άρθρο να λάβουμε υπόψη όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτή την πτυχή θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω και να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να διατυπώσω αυτό το ερώτημα. Ε, πριν από λίγες μέρες αναφέρθηκε ότι η πολιτική αυτή θα περνούσε από την Γενική Επιχείρηση για τις Επιχειρήσεις στη Γενική Διεύθυνση Υγείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτώ, με αυτή τη βάση ποιε θα είναι οι επιπτώσεις, ποια θα είναι η νομική βάση στο τέλος τέλος ε, στην οποία θα βασιστούμε και θέλω να ε, ρωτήσω ποιε θα είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά την έναρξη σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας και εδώ υπάρχουν θέματα αλλαγής νομικής βάσης. Είναι αποσαφηνήσεις που είναι αναγκαίες και πρέπει να τις έχουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω για αυτά τα θέματα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πάρω απαντήσεις. Περνώ στο τρίτο σημείο τώρα. Μετά τον ορισμό των ψευδεπίγραφων προϊόντων, τον καθορισμό της νομικής βάσης που είναι κέρια σημασία στο τρίτο σημείο, οι πωλήσει στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βρίσκεται εκτό τη νομική αλυσίδα δικαιοδοσία τη. Όμω υπαρχουν υπάρχουν κράτη-μέλη όπου η πώληση αυτών των φαρμάκων των σκευασμάτων επιτρέπεται μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτονόητο είναι, είναι σημαντικό να υπάρξει αυτό ο διαχωρισμό. Τι είναι εκτό νομική αλυσίδα και νομική αλληλουχία και τι εντό. Κατά δεύτερον λόγο, πρέπει να μην αφήσουμε εκτό αυτή τη οδηγία αυτό το θέμα το οποίο είναι σημαντικό για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα στην ε, ευρωπαϊκή αγορά μέσω διαδικτύου. Αυτό το θέμα όχι μόνο είναι σημαντικό υπό το πρίσμα του τι αντιπροσωπεύει για την εισαγωγή τέτοιων ε, φαρμάκων ε, που είναι προϊόντα μαϊμούδα στην ευρωπαϊκή αγορά, και πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με τις πωλήσει στο διαδίκτυο. Μια και οι πολίτες, οι κοινοί γνώμοι, έχουν πρόσβαση και πρέπει να, λαμβάνεται να υπόψη είναι αυτό το στοιχείο. Επίσης, αν έχουμε εδώ μπροστά μας το θέμα της ε, παραγωγής προϊόντων απομίμησης, προφανώς πρέπει να γίνει λόγος για ένα τύπο πρακτικής που είναι έγκλημα, εγκληματική πρακτική. Οποιαδήποτε τέτοια πρακτική πρέπει να την χάνει κυρώσεων, να ακολουθούν κυρώσεις ε, σε τέτοιες περιπτώσεις, πρόστιμα, τιμωρίες τι θα γίνει σε σχέση με αυτή, την πτυχή, πώς θα κατηγοριοποιούνται και θα ομαδοποιούνται σε σχέση με τα διάφορα επίπεδα. Εδώ πρέπει να είναι υποχρεωτικές ε, οι διατάξεις για την ασφάλεια, για τέτοια ε, προϊόντα, για φάρμακα. Επίσης, ε, μια συγκεκριμένη κατηγορία των generics πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση που θα κάνουμε παρότι πιστεύω ότι σε αυτή τη διάσταση, στη διάσταση για την ασφάλεια, πρέπει να υπάρξει ένας εναρμονισμός και παρόλα αυτά να μην ξεχνάμε ότι πάντα τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία υιοθετούν τις πιο ενδεδειγμένες διατάξεις ε, και θα μπορούν να ε, υιοθετούν διατάξεις ε, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Είναι θέματα λοιπόν πεπιθήσεων και απόψεων αυτά. Είναι θέματα ε, διατύπωσης ε, και άρθρωσης συμφερόντων που είναι πολλές φορές αντιφατικά μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκόμενων. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια καλή οδηγία που θα επιτρέπει τον συμβιβασμό και αντιστοιχεία αυτών των συμφερόντων με ένα κοινό παρονομαστή ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούμε υπέρ της ασφάλειας της υγείας των ασθενών και την ασφάλιση της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό επανέρχομαι στο θέμα των ορισμών και επανέρχομαι και τονίζω ένα σημείο που είναι σημαντικό για μένα. Η ανάγκη να εντοπίζουμε και να ταυτοποιούμε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα της διανομής φαρμάκων. Υπάρχουν εδώ διάφορες αντιφάσεις όσον αφορά τον κίνδυνο του προϊόντος, τον κίνδυνο της αλυσίδας αυτής οι εμπλεκόμενοι που πρέπει να μας οδηγήσουν στο να διασφαλίσουμε την αλυσίδα περιορίζοντας τους κινδύνους και αυξάνοντας την ασφάλεια. Αυτό θα σήμαινε τη διατήρηση κάποιων ε, διαδικασιών αλλά να μην αφήσουμε εκτός αυτής της διαδικασίας ε, θέματα ασφάλειας και ευθύνης όσον αφορά την αλυσίδα είναι κέρια σημασία εδώ. Όχι μόνο να καθορίσουμε όλους τους εμπλεκόμενους που συμμετέχουν σε αυτή την αλυσίδα, αλλά και να επιμερίσουμε ευθύνε, να καθορίσουμε ποιο είναι ο ρόλος τους, να επιμερίσουμε τις αρμοδιότητες ώστε το κόστος να μην είναι μόνο κάτι το οποίο θα επομίζονται οι καταναλωτές. Είναι απόλυτα αναγκαία αυτή η διαφοροποίηση. Και ζητώ συγγνώμη που ε, το χρησιμοποιώ στα αγγλικά. Ε, μεταξύ traders και brokers ε, ε, η διαφοροποίηση. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό σε σχέση με μια οδηγία που θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, να μπορεί να δημιουργεί μια αλυσίδα διανομής αυτών των ε, φαρμακευτικών προϊόντων που θα είναι αξιόπιστη. Διότι εδώ, σε σχέση με την πιθανότητα εισαγωγής τέτοιων προϊόντων, ψευδεπίγραφων προϊόντων, στην αλυσίδα διανομής, ο κίνδυνος είναι δεδομένος και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να καθοριστούν, να επιμεριστούν ευθύνες, να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος τους, να επιμεριστούν οι ευθύνες και αρμοδιότητες στην αλυσίδα αυτή και να μην υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ε, θα οδηγήσουν να επομίζονται οι καταναλωτές όλα τα κόστη. Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι είναι κέρια σημασίας αφορά το θέμα, το πλαίσιο, το πεδίο της οδηγίας ουσιαστικά όλα τα φάρμακα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την οδηγία. Όλοι οι τύποι και κατηγορίες φαρμάκων και σκευασμάτων, όμως το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Και γι' αυτό σε σχέση με μια θεωρητική προσέγγιση δεν πρέπει να δημιουργούνται προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Μετά από αυτό το σχόλιο θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να έχουμε σαφή διαφοροποίηση και διαχωρισμό μεταξύ των φαρμάκων που αφορούν μία ε, συνταγογράφηση από πλευράς ιατρού και άλλων που δεν υφίστανται υποχρέωση συνταγογράφησης. Αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με τα κράτη-μέλη είναι δεδομένη. Υπάρχουν κράτη-μέλη που διαφοροποιούν και επιβάλλουν ένα τέτοιο ε, καθεστώς προσέγγισης για την ασφάλεια των ασθενών. Μετά από αυτό θέλω να προσθέσω ένα άλλο στοιχείο. Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μια και υπάρχουν φάρμακα εδώ και έχουμε τα generics, θα πρέπει να επιλέξουμε μια ανάλυση κινδύνου. Όμως, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για ψευδεπίγραφο φάρμακο ή απομίμηση φαρμάκου, πρέπει αυτές οι διαδικασίες να ακολουθούνται. Διαδικασίες ασφάλειας, υποχρεωτικές για τα φάρμακα για που ε, υφίστανται στη υποχρέωση συνταγογράφησης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις generics. Μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη σε ισχύ αυτή τη οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μια έκθεση στην Ευρωβουλή με την αξιολόγηση της, ε, ε, των διατάξεων ε, που αφορούν την ασφάλεια. Και έτσι θα μπορούμε να δούμε αν υπάρχει ανάγκη να συμπεριλάβουμε κάτι ή όχι και να ενταχθεί κάτι ή όχι. Και θα μπορούμε να δούμε σε σχέση με την ασφάλεια την συμπερίληψη των φαρμάκων. Αυτή η οδηγία λοιπόν είναι και αναφέρθηκα ότι ο κύριος στόχος είναι η ασφάλεια της υγείας των ασθενών και της δημόσιας υγείας, αφορά όμως και τον έλεγχο των, της ποιότητας των εισαγόμενων προϊόντων. Εδώ είναι που ανοίγει πόρτα και παράθυρο για την εισαγωγή τέτοιων ψευδεπίγραφων προϊόντων μαϊμούδων. Εδώ πρέπει λοιπόν με βάση τη διεθνή συνεργασία να προσπαθήσουμε με τις βέλτιστες πρακτικές να ακολουθήσουμε τη σωστή πορεία. Μόνο ένα σχόλιο ακόμα και ολοκληρώνω. Μια τελευταία παρατήρηση που αφορά το πλαίσιο, το πεδίο της οδηγίας και που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να το συμπεριλάβουμε όσον αφορά την, ε, ε, διάταξη, στη διάταξη αυτή για τα φάρμακα. Ολοκληρώνω όπως ξεκίνησα, Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μια οδηγία που θα αρθρώνει και θα βρίσκει ένα κοινό παρονομαστή μεταξύ των αντικρουόμενων συμφερόντων. Αυτός ο κοινό παρονομαστής ως στοιχείο είναι η ασφάλεια της υγείας των ασθενών και της δημόσιας υγείας. Ολοκληρώνω και επαρκούμε σε αυτά που είπε. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σχόλια και παρατηρήσεις που έχουν να υποβάλουν οι συνάδελφοι, οι σκιώδεις εισηγητές σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή, μια κοινή πορεία μεταξύ αντικρουόμενων στοιχείων μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ολοκληρώσω και μια κοινή πρώτη φορά που υποβάλλω μια πρόταση έκθεσης μέσα σε αυτή την Επιτροπή Θέλω να ευχαριστήσω την εξαιρετική εργασία και την υποστήριξη τεχνική που δόθηκε σε μένα από πλευράς της πολιτικής ομάδας και γραμματείας και θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την υποστήριξη. Είναι μεγάλη η ευθύνη που αναλαμβάνουν και έτσι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία αλλά η ευθύνη φυσικά για την έκθεση είναι δική μου και πρέπει να δραχθούμε τι ευκαιρίες για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, σε μια πρόταση που θα διασφαλίζει την υγεία και τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Συγήτρια, για τη δουλειά σας, την οποία σίγουρα εκτιμούν οι συνάδελφοι. Η κυρία Γκόστετ είναι η πρώτη που ζητάει τον λόγο στα πλαίσια της συζήτησης που ακολουθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς την εισηγήτρια για την προσπάθειά της μέχρι σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η έκθεση, αυτή την οδηγία, την περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και χρόνια την απαιτούσαμε και τη ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πραγματικά υπάρχει κίνδυνος εδώ, σε ό,τι αφορά τους ασθενείς. Εγώ θεωρούσα ανέκαθεν ότι η απομίμηση φαρμάκων ισοδυναμεί με έγκλημα. Γιατί ξέρουμε ότι ένα ψευδεπίγραφο φάρμακο στην καλύτερη περίπτωση δεν θεραπεύει και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να είναι εξαιρετικά βλαβερό. Για να μην πω εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία, μπορεί να προκαλέσει μάλιστα και το θάνατο. Η συγγήτρια μας είπε ότι αφορούσε το 10% του κύκλου εργασιών της ε, φαρμακοβιομηχανίας είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ το κέρδη από τα ψευδεπίραφα φάρμακα. Υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά που ανέφερε η συγγήτρια, θα ήθελα να υπογραμμίσω πολύ γρήγορα κάποια σημαντικά σημεία. Καταρχάς, συμφωνώ με την έκθεση για τη διπλή νομική βάση. Συμφωνώ να υπάρχει ένας ε, πολύ ευρύς ορισμός του ψευδεπίγραφου φαρμάκου, δηλαδή αυτός ο ευρύς ορισμός, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αφορά και τα φάρμακα που συνταγογραφούνται, καθώς και αυτά που είναι εκτός συνταγογράφησης, καθώς και τα γενώσιμα φάρμακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή ε, θα έχουμε μια νομοθεσία αυστηρή για κάποια είδη φαρμάκων, ενώ κάποια άλλα εκφεύγουν αυτού του πλαισίου. Αν τα φάρμακα είναι παραποιημένα, γενώσιμα ή όχι, συνταγογραφούμενα ή όχι, αν είναι ψευδεπίγραφα, είναι αυστηρά, ε, είναι σαφώς ε, επικίνδυνα για τους ασθενείς. Θέλω λοιπόν ε, μια ευρία νομοθεσία και έναν ευρύ ορισμό. Το επιχείρημα ότι δεν έχει νόημα για φθηνά φάρμακα γενώσιμα να εφαρμόσουμε την νομοθεσία, αυτό το επιχείρημα για μένα δεν είναι βάσιμο. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ταυτότητα του φαρμάκου. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί αν θέλουμε να γενικεύσουμε ένα σύστημα προστασίας ενιαίο στα 27 κράτη-μέλη και αυτό το σύστημα προστασίας να είναι συμβατό ε, στις διάφορες χώρες, το τίμημα ή μάλλον ε, η τιμή θα μειωθεί χάρη σε αυτές τις οικονομίες κλίμακας. Αν υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο προστασίας, νομίζω ότι αποδυναμώνουμε την ασφάλεια της αλυσίδας ανεφοδιασμού και τότε θα υπάρχει επιπλέον κόστος. Αν έχουμε μια αυστηρή νομοθεσία για το σύνολο των φαρμάκων, στο σύνολο των 27 κρατών μελών, τότε ε, μειώνουμε προφανώς το κόστος ε, του αγώνα καταπολέμησης των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Κάτι άλλο που μου φαίνεται σημαντικό είναι η απαγόρευση της ανασυσκευασίας, της νέας συσκευασίας. Αν θέλουμε να αποφύγουμε και να μην δώσουμε τη δυνατότητα απομίμησης του φαρμάκου, θα πρέπει να απαγορεύσουμε κάτι τέτοιο, αυτή την ε, πρακτική. Είναι ο πρώτος κανόνας αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την ε, απομίμηση του φαρμάκου. Θα πρέπει μεταξύ του εργαστηρίου, δηλαδή που παρασκευάζει το φάρμακο και του ασθενούς, κανένας, κανένας ενδιάμεσος, κανένας μεσάζοντας να μην έχει το δικαίωμα να ανοίξει το κουτί με το φάρμακο. Αυτό είναι στοιχειώδες για κάτι την απόψή μου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μιλήσω στεναρά ε, ότι πρέπει να απαγορεύεται να ανοίγουμε το κουτί και να ανασυσκευάζουμε το φάρμακο. Αυτό είναι θέμα εμπιστοσύνη και λογική μου φαίνεται. Τώρα, ποια λύση θα προτείνουμε. Με την ταυτότητα του φαρμάκου φυσικά θα έχουμε ε, γραμμικούς που θα ταυτοποιούν το φάρμακο. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Να μην ανοίγουμε το αρχικό κουτί του φαρμάκου, γιατί σας είπα ότι δεν θέλω να το ανοίγουμε αυτό το αρχικό κουτί, αλλά θα βάλουμε ένα νέο κουτί εξωτερικό, το οποίο θα ε, σέβεται τις απαιτήσει του κράτους μέλους εισαγωγής. Γιατί ξέρουμε το φάρμακο κυκλοφορεί από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Και θα πρέπει πάνω στην, στο κουτί να υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον ασθενή. Στη γλώσσα της χώρας του. Στη χώρα δηλαδή του κράτους εισαγωγής του, ώστε ο ασθενής να ενημερώνεται σωστά. Δύο κουτιά λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων στην αλυσίδα νεφοδιασμού αυτοί οι εμπλεκόμενοι είναι πολύ άριθμοι. Υπάρχει ο κατασκευαστής, υπάρχουν τα άτομα τα οποία μπορούν να διανέμουν τα φάρμακα, υπάρχουν οι έμποροι, ε, υπάρχουν οι φαρμακοποιοί. Επίσης, η κατανομή ευθυνών σε όλους τους ε, εμπλεκόμενους που δραστηριοποιούνται σε αυτή την αλυσίδα και προμηθεύουν το φάρμακο, ε, θα πρέπει να καθοριστεί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπόκειται σε επιθεωρήσεις και το είπε και η συγγήτρια ούτως ή άλλως, ανάλογα με, την, με τους κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να επικαιροποιούνται και λαμβάνοντας υπόψη το πώς έχουν λάβει ο καθένας την αδειά του. Θα πρέπει ο έλεγχος να γίνεται επιπλέον πέρα από τις επιθεωρήσεις, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία. Και νομίζω ότι το ανέφερε και αυτό η συγγήτρια. Τέλος, τελειώνω με ένα σημείο που μου φαίνεται επίσης πολύ σημαντικό είναι το ίντερνετ. Συνηθίζω να λέω ότι σε ό,τι αφορά την απομίμηση των φαρμάκων, καλύτερα να ενημερώσουμε τον ασθενή ότι δεν θα πρέπει να αγοράζει φάρμακα στο ίντερνετ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα περισσότερα φάρμακα που πουλούνται στο ίντερνετ είναι ψευδεπίγραφα. Προσοχή λοιπόν ε, στην διαφήμιση στις ε, μηχανές αναζήτησης προσοχή στα φαρμακεία που είναι online και που δεν έχουν άδειε. Θα πρέπει να κάνουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ε, των καταναλωτών, των χρηστών του ίντερνετ για τους κινδύνους αγοράς των φαρμάκων online. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Νομίζω ότι θα πρέπει να προλάβουμε αντί να διορθώσουμε. Θα πρέπει να προβλέψουμε ένα κανονισμό ή μια ειδική οδηγία για το εμπόριο online. Αυτά προς το παρόν, κυρία Πρόεδρε, για αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Γκοστέτ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μπέρεντ, θα ήθελα να σας πω ότι μια φλαμανδική, ένα φλαμανδικό κανάλι θέλει να κινηματογραφήσει τον κύριο Κλάς. Έχει κανένα αντίρρηση? Όχι. Πολύ ωραία. Η κυρία Μπέρεντ Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από την εισηγήτρια ότι καθυστέρησα και έφτασα όταν είχε αρχίσει την παρέμβασή της. Μου είχαν πει ότι στις 10.30 θα ξεκινούσαμε. Και αυτό δεν κάνει τα πράγματα απλούστερα, ούτε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θέλουμε να συζητούμε τι παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Λαλίση ήρθε εδώ ασθμένουσα. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αλλά για τις ικανότητες για να δουλέψουμε αποτελεσματικά και για να είμαστε σοβαροί, παρακαλώ στο Προεδρείο να συζητηθεί αυτό. Όταν θα έχουμε συζήτηση θεμάτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τότε <clears throat> είναι λογικό να τηρούμε τις χρονικές ενδείξεις του προγραμματισμού, του σχεδιασμού. Λυπούμε. Έφυγα και από άλλη συνεδρίαση και γι' αυτό καθυστέρησα να φτάσω εδώ. Κυρία Πρόεδρε τώρα, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που ήδη προηγούμενα όταν συζητήσαμε την έκθεση είχα κάνει και ήδη και σε συζήτηση με την εισηγήτρα είχα αναφέρει κάποιες παρατηρήσεις. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ε, έκθεση από πλευρά τη. Δεν είναι εύκολο όταν αναλαμβάνει κανεί τη σύνταξη έκθεση για πρώτη φορά με ένα τέτοιο περίπλοκο θέμα. Συγχαίρω την κυρία Ματίας που τα κατάφερε πραγματικά για το έργο που επετέλεσε, που είναι εξαιρετικό, και την ταχύτητα και το βάθος στο οποίο εργάστηκε για αυτό το θέμα. Γι' αυτό είναι και εύκολο για μένα να πω ότι σε πολλά σημεία συμφωνώ απόλυτα μαζί τη Εκεί στις ε, απόψεις που διατυπώνει. Πιστεύω ότι και πολύ καλά για την νομική βάση για το άρθρο 95 και το 152 άρθρο μπορεί να προσθεθεί. Αυτό δεν βλάπτει. Ίσα ίσα την επικέντρωση της πολιτικής μας για τη δημόσια υγεία την διασφαλίζει, το είπε και η κυρία Γκροστέτ, συμφωνώ μαζί της. Πιστεύω επίσης όπως και η κυρία Ματίας και όπως και η κυρία Γκροστέτ και εγώ, πιστεύω ότι η επικέντρωση αυτών που κάνουμε εδώ πρέπει να είναι η ασφάλεια, η νομική ασφάλεια υπέρ των, ασφαλών, πρέπει να, ε, ασθενών. Πρέπει να προστατεύονται οι ασθενείς είτε εναντί φαρμάκων που χρησιμοποιούν χωρίς να έχουν το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμείτε παίρνουν ένα ας το πω έτσι ε, ορμονικό ε, προϊόν ή ένα σκεύασμα κατά του καρκίνου που ελπίζουν ότι θα προστατευτούν από την ασθένειά τους όμως ε, δεν έχουν κάποια αποτελεσματικότητα ή δεν είναι καθαρά όσον αφορά τη σύστασή τους είναι και δεν έχουν παραχθεί με ασφάλεια. Η ασφάλεια των ασθενών είναι η κύρια λοιπόν σκέψη που πρέπει να πριτανεύει στο έργο μα. Συμφωνώ απόλυτα με τη Μαρίζα Ματιάς και την κυρία Γκροστέτ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Γι' αυτό ο ορισμός πράγματι είναι ουσιοδέστατο στοιχείο και πολλοί άλλοι τομεί ε, που αναφέρθηκαν από τις δύο κυρίες αληθεύουν. Πρώτα για τον ορισμό λοιπόν. Πολύ συχνά συμφωνώ απόλυτα με την Φρανσουάζ Γκροστέτ, παρότι ανήκουμε και σε διαφορετικά κόμματα, όμως εδώ δεν συμφωνώ και όπως η κυρία Ματίας ξεκίνησε και είπε, εδώ πρέπει να πω ότι για την ασφάλεια όσον αφορά τα προϊόντα απομίμησης πρέπει να ξεκινήσουμε με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Πρέπει γι' αυτό τον λόγο να ξεκινήσουμε με τα υποσυνταγογράφηση φάρμακα, γιατί είναι διαφορά μεταξύ ενός φαρμάκου που έχει υποχρέωση συνταγογράφησης και ενός άλλου που δεν έχει τέτοια ε, υποχρέωση. Η ιδιότητα για τα υποσυνταγογράφηση φάρμακα είναι ότι εν δυνάμει μπορεί να έχουν τέτοιες επιπτώσεις και ε, επιπτώσεις στον ασθενή που μόνο ένας ε, γιατρός μπορεί να το συνταγογράψει. Αυτά τα οποία μπορούν να απολυθούν σε ένα φαρμακείο όσον αφορά την αυτοφαρμακευτική θεραπεία δεν εντάσσονται μέσα στην ε, θεραπεία από τον ιατρό και παρακολούθηση από τον ιατρό. Αν καταφέρουμε να έχουμε ένα στεγανό, ασφαλέστατο σύστημα, πολύ ωραία τότε όπως είπε η κυρία Ματιάς μετά από πέντε χρόνια να το ξαναδούμε και να το διευρύνουμε το εύρος. Όμως αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ασθενείς είναι από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και όχι φάρμακα lifestyle ή άλλα που πολλούνται στο διαδίκτυο. Σε αυτό θα έρθω σε ένα λεπτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι η επικέντρωση όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα ορθή επικέντρωση. Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα πρώτα πρέπει να καλύπτονται. Τι θα κάνουμε με το safety feature. Έχει κάνει κάποιες προτάσεις η κυρία Μάτιας. Πιστεύω ότι είναι σωστό να έχουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση, σαφή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η κυρία Γκροστέ τι είπε. Είπε κάτι γι' αυτό ότι μέσω της απαγόρευσης της ανασυσκευασίας πρέπει να προχωρήσουμε. Μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Αλλά αυτό θα είναι υποψία ότι θέλουμε το παράλληλο εμπόριο να βλάψουμε. Μου είναι αδιάφορο το θέμα των παράλληλων εμπόρων. Εκείνο που δεν μου είναι αδιάφορο είναι το θέμα της υγείας των ασθενών, οι ασθενείς. Γι' αυτό μου είναι αδιάφορο. Αν θα έχουμε ένα overboxing, ανασυσκευασία, η δεύτερη συσκευασία. Αν το επιτρέψουμε αυτό, Φρανσουάζ, θα πρέπει στο overbox να έχουμε τα θέμα safety features. Γιατί με την ανάγνωση από το φαρμακείο με ηλεκτρονικό τρόπο, το scanning, δίνει την ικανότητα να ανοιχνεύεται ότι είναι ασφαλές από το, τη συσκευασία. Εκείνο που θέλω όμως οπωσδήποτε να απαγορευτεί είναι η σημερινή, πώς να το πω, πρακτική. Ότι για παράδειγμα, πακέτα φαρμάκων μπορούν να ε, αποκόπτονται. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αποκοπή από, τους, από τη συσκευασία ε, σε κομμάτια των επιμέρους συσκευασμάτων. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να απαγορεύεται. Αν, για παράδειγμα, εγώ πρέπει να ανοίξω το, τη συσκευασία, τη συσκευασία του φαρμάκου μου και μου πέσουν δύο ε, συσκευασίες, ε, μια των 10 και μία των 5 ή σε διαφορετική ομαδοποίηση πέφτουν τα φάρμακα, αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό οι μονάδες ε, στις οποίες πολλούνται αυτά θα πρέπει να εξετάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των ασθενών. Θέλω να ρωτήσω εν τέλει αν τα generics πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά τα γενώσιμα και εδώ πάλι πρέπει να πω, συμφωνώ με όλους εκείνους και νομίζω και με την εισηγήτρια μπορώ να πω, που λένε ότι αν έχουμε ένα ψευδεπίγραφο και έχουμε ένα γενώσιμο το οποίο εξακολουθεί να είναι υπόχρεο προς συνταγογράφηση. Μου είναι αδιάφορο αν αυτό το φάρμακο τώρα είναι αρχέτυπο χύψη ή ε, ε, ωμέγα ή ένα οποιοδήποτε άλλο από πλευράς ονομασίας. Από πλευράς της συνταγογράφησης και παρακολούθησης του γιατρού ίσως ε, τα προϊόντα αυτά είναι λιγότερο, ας το πω έτσι, κερδοφόρα στην απομίμηση. Αν δει κανείς όμως τι έχει γίνει στο παρελθόν με προϊόντα απομίμησης, με προϊόντα μαϊμούδες, ίσως αυτό το επιχείρημα δεν στέκει. Όμως, στον ορισμό θα πρέπει η παρακολούθηση με τον γιατρό να είναι το σημείο αναφοράς, η συνταγογράφηση δηλαδή. Τότε είναι αδιάφορο αν το ένα προϊόν είναι αρχέτυπο ή το άλλο είναι γενώσιμο. Λοιπόν, αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τώρα, το θέμα του εμπορίου στο διαδίκτυο. Όλοι συμφωνούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι το ε, εμπόριο στο διαδίκτυο. Αν καταφέρουμε εδώ να έχουμε ε, κάτι το οποίο θα ε, μεγεθύνει την ασφάλεια, θα επαυξήσει την ασφάλεια, θα είναι εξαιρετικό. Για παράδειγμα, όσον αφορά <clears throat> την συνταγογράφηση, την εγγραφή στο, σε, σε συνταγή γιατρού, να υπάρχει η δυνατότητα μόνο με labor μέσω του διαδικτύου ή μέσω ενός λογότυπου που θα διασφαλίζει την χρήση ενός φαρμάκου ή ενός, ε, την πώληση μέσω ενός φαρμακείου στο διαδίκτυο. Quality labor for e-pharmacies για την ηλεκτρονική εμπορία μέσω φαρμακείων στο διαδίκτυο. Θα πρέπει δηλαδή να μην αναγκάζεται κανείς να χρησιμοποιεί μια ε, ιστοσελίδα αμερικανική, αλλά μια ιστοσελίδα που θα έχει σαφές labeling, που θα δείχνει ότι υπάρχει νομιμότητα. Δεν θα εξαφανίζεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Αν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό ως πρότυπο, θα είναι πρότυπο και για τους άλλους στο διαδίκτυο και για την πιστοποίηση και αδειοδότηση και σε άλλες ιστοσελίδες ή σε άλλες δυνατότητες πώλησης ε, στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήθελα απλώ να σα πω ότι ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί χθε τροποποιήσαμε την ημερήσια διάταξη και δεν ε, συζητήσαμε ένα από τα σημεία και γι' αυτό συζητήθηκε νωρίτερα αυτό το σημείο. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Τρεμόπουλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω την απόφαση της Επιτροπής να μεταφέρει τις αρμοδιότητες για τα θέματα των φαρμάκων και των φαρμακευτικών οργάνων από τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή. Αυτό ήταν ένα αίτημα της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίξαμε και εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα των Πράσινων καθώς και ένα ζήτημα δημόσιες υγείας ε, που έπρεπε να ρυθμίζεται με βάση τα κριτήρια ε, αυτών ε, που πρέπει να ελέγχουν και όχι των συμφερόντων της φαρμακοβιομηχανίας. Το έχω πει και στην αίθουσα αυτή. Θα πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει και αυτό που ο Ιπποκράτης έχει πει ε, ότι η τροφή σου είναι το φάρμακό σου και να προσθέσω ότι η υγεία της φύσης είναι και η υγεία των ανθρώπων. Τώρα βέβαια έχουμε ε, διαδεδομένη χρήση φαρμάκων που καταπολεμούν το σύμπτωμα και όχι την ίδια την αιτία. Με πολύ μεγαλύτερη απειλή της δημόσιας υγείας αποτελούν και τα ψευδεπίγραφα φάρμακα που συζητάμε και τα οποία είναι σαφές ότι δεν θέλουμε να εισάγονται αλλά ούτε και να εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περιμένουμε την ε, γραπτή έκθεση της συγγήτριας... όμως μπορούμε να πούμε από τώρα ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι σε καλή κατεύθυνση και ένα απαραίτητο βήμα για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Θα ήθελα όμως να μείνω σε κάποια σημεία, κάποια ήδη αναφέρθηκαν, πιστεύω να το δούμε το θέμα πιο προσεκτικά Καταρχάς η επιχειρηματολογία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα δεν πρέπει να αναλωθεί σε συζητήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, το παράλληλο εμπόριο ή ακόμη και τα αντίγραφα φάρμακα, καθώς αυτά αφορούν κυρίως εμπορικές διαστάσεις του ζητήματος και όχι τόσο προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Δεύτερον, πρέπει να εισάγουμε ρυθμίσεις για να καταπολεμήσουμε τις παράνομες διαδικτυακές πωλήσει, που είναι η κύρια πηγή των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Η πρόταση της Επιτροπής ασχολείται μόνο με την ε, παραδοσιακή αλυσίδα διανομής ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά, ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για να καταπολεμήσουμε τις παράνομες διαδικτυακές πωλήσει, έστω και αν από νομική πλευρά η οδηγία δεν μπορεί να εισάγει άμεσε ρυθμίσει για διαδικτυακά φαρμακεία και παράνομες πωλήσει. Μπορούν παρόλα αυτά να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, όπως η απαγόρευση πληρωμένων διαδικτυακών καταχωρήσεων που οδηγούν σε παράνομα διαδικτυακά φαρμακεία. Η δημιουργία ενός διαδικτυακού μητρώου πιστοποιημένων διαδικτυακών φαρμακείων σε χώρες, σε εκείνες τις χώρες όπου επιτρέπεται η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων. Καθώς και η δημιουργία ενιαίου λογότυπου πιστοποίησης διαδικτυακών φαρμακείων. Τρίτον, πρέπει να υπάρξει ένας πιο ξεκάθαρος ορισμός για το τι είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Με βάση τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του Δεκεμβρίου του 2008. Ούτως ώστε να διατηρήσουμε συμπαγή τη διεθνή συνεργασία των κρατών μελών. Τέταρτο, χαιρετίζω την πρόθεση της Επιτροπής για ενδυνάμωση των ελέγχων όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα διανομής, όπως επίσης και όλων των ενεργών συστατικών. Θα ήθελα να μεταφέρω το αίτημα για υποχρεωτική εγγραφή σε Μητρό όλων των εμπλεκόμενων στην νόμιμη αλυσίδα προσφοράς, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο και θα είναι διαθέσιμο στο κοινό. Τέλος, να πω ότι πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει συνεχής και ξεκάθαρη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού για να κάνει ενημερωμένες και υπεύθυνες αγορές καθώς και για να συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό και την αναφορά των παράνομων ενεργειών και φαρμάκων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Κυρία Μαρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω ότι ε, συμφωνώ με σχεδόν όλα από αυτά που ανέφερε η συγκήτρια εκτός από ένα σημείο. Αν κάτι πάει στραβά δεν φταίει εκείνη, φταίμε όλοι γιατί ήταν ομαδική η δουλειά που κάναμε. Στους ε, ορισμούς και το τι πρέπει να κάνουμε. Θα ήθελα να πω τα εξή. Για το αν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα συνταγογραφούμενα, τα μη συνταγογραφούμενα, τα γενώσιμα ή όχι κλπ. Εγώ νομίζω ότι αν επηρεάζει δυσμενώ τον ασθενή, είναι καθήκον μα να το εξετάσουμε. Υπάρχουν δύο τομείς που πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και που νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε στο παρόν στάδιο. Καταρχήν, η οδηγία πρέπει να είναι εφικτό να μπορούμε να τη διαχειριστούμε, να εξετάσουμε τα θέματα της συσκευασία, τα θέματα της διανομής ε, και όλα αυτά και ο τόπος διανομής είναι μια πρόκληση γιατί μερικές φορές ε, προέρχονται από μικρά φαρμακεία και γι' αυτό θέλουμε ε, να μην δημιουργήσουμε και δυσμενείς ε, οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή θέλουμε να προστατεύουμε τους ασθενείς ε, και παράλληλα να έχουμε κάτι το οποίο να μπορούν και οι επιχειρήσεις να αποδέχονται και να μπορούν να δουλέψουν με αυτό. Για το θέμα του διαδικτύου, ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα που συνεχώς αλλάζει και αυτό το οποίο τώρα συζητάμε μπορεί να αλλάξει σε λίγα χρόνια. Από όσο γνωρίζω, το 50% των ψευδεπίγραφων φαρμάκων προέρχεται από το διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το διαδίκτυο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι όμω το οποίο τροποποιείται συνεχώ και πρέπει συνεχώ να είμαστε σε γρήγορση ώστε να λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία θα προκύψουν. Το να βάλουμε ένα λογότυπο δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει γιατί μπορεί εύκολα να αντιγραφεί. Να το εξετάσουμε πάντως. Euh, Ο κύριος Πέτερ Λίζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ματίας. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλή η πρόταση την οποία έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα. Υπάρχουν τα θέματα, του, καταρχήν το ότι είναι επίγον να αντιμετωπίσουμε τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στον ασθενή. Επίσης, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται η συζήτηση το ότι αν ε, προχωρήσουμε υπερβολικά μπορεί να διαταράξουμε τις ε, παράλληλες εισαγωγές και πρέπει να δούμε και το θέμα των παράλληλων εισαγωγών. Και το πρόβλημα είναι ότι αν δεν έχουμε παράλληλες εισαγωγές μπορεί σε ορισμένες χώρες να αυξηθεί το κόστος των φαρμάκων που μπορεί να πει κανεί ότι πρέπει να καταβληθεί αυτό το επιπλέον κόστο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και την πολιτική πραγματικότητα. Ότι μιλάμε για το συμφέρον των ασθενών και δεν είναι προ συμφέρον των ασθενών να αυξάνεται το κόστο των φαρμάκων. Και παίζει ρόλο και η τιμή του φαρμάκου στο τι χρηματοδοτείται από το Δημόσιο Σύστημα Υγεία, παραδείγματο χάρη. Ε, ιδανικό θα ήταν σε έναν τέλειο κόσμο να έχουμε παράλληλε εισαγωγέ με τι ίδιε τιμέ δεν θέλουμε ε, να έχουμε τέτοια διαφορετικά συστήματα στην Ευρώπη. Καλό θα ήταν να είχαμε μία νέα τιμή φαρμάκου, αλλά οποιοδήποτε ασχολείται με αυτό το θέμα ε, σίγουρα γνωρίζει ότι δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να επιληθεί μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν συζητήθηκε το θέμα και προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία και ε, υπέρ της ασφάλειας και με την τήρηση των παράλληλων εισαγωγών. Όσον αφορά την επιτροπολογία, ε, βλέπουμε σχετικά συχνά μέσα στην πρόταση ότι η Επιτροπή αποφασίζει, η Επιτροπή κάνει κλπ. Ενώ εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέλαμε ε, να γνωρίζουμε επακριβώ τι σημαίνει όταν αποφασίζουμε κάτι. Δεν θέλουμε να δώσουμε λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό νομίζω αξίζει τον κόπο να περιγράφουμε λίγο πιο συγκεκριμένα το τι κάνουν οι παραγωγοί φαρμάκων και τι κάνει ο κάθε εμπλεκόμενος στην αλυσίδα και τι ε, κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Να μην τα αφήσουμε όλα δηλαδή στην επιτροπολογία και στη διαδικασία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα πρέπει επίσης ε, να φροντίσουμε και την ασφάλεια αλλά και την προστασία των δεδομένων. Ε, γιατί ε, υπάρχει κίνδυνος διαρροής πληροφοριών αν υπάρχει ε, αλλαγή συσκευασία. και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Να δούμε αν το φάρμακο φτάνει στη μορφή ε, που το, στην οποία το παρασκεύασε ο κατασκευαστής, αν φτάνει στη μορφή αυτή και στον ασθενή. Υπάρχουν θέματα τα οποία τα γνωρίζουν οι αρχές επιτήρησης που δεν μπορεί να τα γνωρίζει ο καταναλωτής και επομένως είναι σημαντικό να προστατεύσουμε και τα προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορεί ο κατασκευαστή να γνωρίζει ποιο ασθενή θα πάρει το φάρμακο, γιατί υπάρχουν προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να, να διαραίουν. Όσον αφορά το διαδίκτυο, υποστηρίζω όλα αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε και στο κείμενο αυτό να ασχοληθούμε με τους κινδύνους που προέρχονται από το διαδίκτυο. Όσον αφορά το overboxing, το να τοποθετεί ένα κουτί πάνω από το αρχικό κουτί, είναι ένα θέμα προς συζήτηση, νομίζω το έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως και στο θέμα των τιμών έχουμε το πρόβλημα ότι δεν, μπορούμε να έχουμε, δεν έχουμε ένα αρμονισμένο σύστημα και μεγέθη συσκευασίας και εφόσον ισχύει το τωρινό σύστημα, δεν λύνεται με το overboxing το πρόβλημα. Έχω λοιπόν και εδώ ένα ερωτηματικό για το κατά πόσο είναι εφικτό το σύστημα του overboxing. Γιατί ε, διπλή νομική βάση, ξέρουμε τα σχετικά με το άρθρο 152 και από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αν ε, σωστά έχω καταλάβει, θα πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένα σε ποιο άρθρο αναφέρεται η νομική βάση. Δεν μπορούμε να πούμε θα έχουμε τη διπλή νομική βάση για να βοηθήσουμε σε θέματα υγείας. Δεν είναι απλό από νομικής πλευράς. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ποιες περιπτώσεις εμπίκνουν στο 152 και σε ποιες το άρθρο 192. Ανέφεραν αρκετοί συνάδελφοι ότι η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνη για τα θέματα ανταγωνισμού τώρα και ε, συμφωνώ όλο αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα πρέπει να έχουμε το άρθρο 152 ως βάση γιατί επί χρόνια οι προτάσεις που γίνονται στα θέματα του περιβάλλοντος μπορεί να προέρχονταν και, με βάση το, και, και από το άρθρο 192. Προβλέπεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ε, υγείας και δεν χρειάζεται κάθε φορά να έχουμε διπλή νομική βάση και στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα της υγείας. Μπορούμε να δουλέψουμε και με το άρθρο 192 σαν νομική βάση ανεξάρτητα από ποια γενική διεύθυνση προέρχεται το θέμα. Βέβαια δεν έχω αντίρρηση Απλώς ε, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευκρινείς σε αυτά τα οποία προτείνουμε. Και θέτω ε, την ερώτηση και προς την Επιτροπή ε, τι προβλέπει σχετικά με την νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Κύριε Παρβάνοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. <clears throat> Και εγώ συγχαίρω την Κομισιόν για το πολύ φιλόδοξο σχέδιο αυτό, την πολύ φιλόδοξη πρόταση, γιατί τη ζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και επιτέλους ήρθε. Συγχαίρω επίσης την εισηγήτρια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί συνένεση για τα θέματα της πρότασης. Παρότι, από ό,τι φαίνεται, συγκλίνουμε προς αυτό τώρα. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Ορισμένες ε, σχετίζονται με την ε, ε, έκθεση που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελέτη και που είναι η μελέτη αντικτύπου για την νόμιμη και παράνομη αγορά φαρμάκων, καθώς και τα δεδομένα με τα οποία κάνουμε τις εκτιμήσεις μας. Μια έννοια που πρέπει να συζητηθεί είναι η επίπτωση των μέτρων στις τιμές των φαρμάκων για τους ασθενείς και για τους καταναλωτές. Ε, στην έκθεση η Κομισιόν λέει ότι ο κλάδος ε, μπορεί να αντισταθμίσει και να απορροφήσει το, την επίπτωση όλων των νέων μέτρων, παρότι δεν μας επιβεβαίωσε ο κλάδος όλες τις συναντήσεις που είχαμε κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά το ακούμε. Ακούμε ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει, να απορροφήσει αυτό το κόστος. Επίσης, ε, σε καμία περίπτωση θα πρέπει ο ασθενής ή η καταναλωτής να φέρει το κόστος. Θα ήθελα να έχουμε μία μελέτη για την εφαρμογή των μέτρων. Ε, συνήθως ε, την έκθεση αυτή την έχουμε πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ. Αλλά μια και το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό ε, και επειδή μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στι τιμέ των φαρμάκων, καλό θα ήταν να έχουμε αυτή την έκθεση τρία χρόνια μετά για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, καθώ και την ανάγκη ενδεχομένω να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε τα κριτήρια για την ανιχνευσιμότητα, τη βάση των κριτηρίων και αν θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα προϊόντα. Παραδείγματο χάρη τα γενώσιμα, τα οποία δεν τα παραπεί κανεί, δεν τα απομιμείται. Αν αυτά τα μέτρα θα αφορούν όλα τα φάρμακα, προφανώ θα επηρεάσουν σημαντικά όλη την αγορά. Παρότι το, μόνο το 0,7% των γενώσιμων ε, παραπείται. Επίσης, για το διαδίκτυο. Ε, προσοχή να μην ε, υπάρχουν, υπάρξουν προβλήματα ιδιωτικής σφαίρας. Παραδείγματο χάρη το είδος ε, των φαρμάκων που πουλάει ένα φαρμακείο, καθώς και την ποσότητα των φαρμάκων, δεν θα πρέπει αυτές τις πληροφορίες να τις έχει ο κατασκευαστής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε το σύστημα τι θα καλύπτει σε ό,τι αφορά την ανιχνευσιμότητα. Η πρόταση αυτή δεν αντιμετωπίζει το θέμα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων 100%. Ε, οι συνάδελφοι είπαν ότι μόνο ένα ποσοστό αντιμετωπίζει των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Επίσης θα πρέπει να δούμε το θέμα του ίντερνετ, γιατί γίνονται μεγάλες πωλήσει φαρμάκων από το ίντερνετ, το ξέρουμε, και η πρόταση αυτή δεν καλύπτει αυτό το σημαντικό θέμα. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ για αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι με αυτό το νομοθέτημα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα με τα φάρμακα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να ζητήσουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της Κομισιόν ε, και επίσης να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για τους κινδύνους αγοράς, πώλησης και αγοράς φαρμάκων από το ίντερνετ. Για μένα η ε, απομίμηση είναι οργανωμένο έγκλημα, απομίμηση φαρμάκων. Έχουμε τη γνωμοδότηση του ΠΟΕ. Για τα ποσοστά των ε, φαρμάκων που, που απομιμούν, παραποιούνται συγγνώμη, ε, μέσα από τα νόμιμα κυκλώματα, το ποσοστό αυτό είναι μικρό. Επίσης, θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν και το Συμβούλιο τι πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε ε, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό ε, στο πρίσμα της ε, αστυνομικής συνεργασίας. Τώρα θα ήθελα να διαβάσω κάτι στα βουλγαρικά. Δεν έχω. Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα είναι απειλή που δεν, αφορά, που δεν είναι μόνο οργανωμένο έγκλημα, αλλά είναι έγκλημα κατά της δημόσιας υγείας. Η Κομισιόν είναι πολύ ευαίσθητη για αυτό το θέμα και προσπαθεί να ανταποκριθεί ε, όχι μόνο με νομοθετήματα, αλλά και με επιχειρησιακούς τρόπους, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των ε, σχετικών και αρμοδίων αρχών. Προβλέπονται επίσης κάποιες κυρώσεις, καθώς και διοικητική συνεργασία με τους κατασκευαστές. Επίσης θα πρέπει να προβούμε και στη λήψη κατασταλτικών μέτρων. Πρέπει να δούμε πώς θα διοδοτούνται τα φάρμακα. Θα θέλαμε ε, η Κομισιόν να αντιμετωπίσει το, την παράνομη πώληση και να αντιμετωπίσει την ε, πώληση ψευδεπίδαχων φαρμάκων ως οργανωμένο έγκλημα. Θα ήθελα να δοθεί συνέχεια σε αυτό το θέμα. Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί ε, σοβαρά και το κακό θα πανταχθεί στη ρίζα του. Ευχαριστώ και ο Σίμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης την εισηγήτρια παρότι είναι καινούρια πολύ καλά διατυπώνει τις σκέψεις της, έκανε πολύ καλή δουλειά. Αυτή η έκθεση δείχνει και η συζήτηση δείχνει ότι η πολιτική ακολουθεί, χωλαίνει πίσω από την πραγματικότητα. Θα πρέπει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο να τα δούμε αυτά. Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για την πολιτική υγεία σε επιτραπέζεις. Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο ανοίγει νέε δυνατότητες για τους ασθενείς και ότι αλλάζουν οι συνθήκες ε, εμπορίας και της αγοράς. Με αυτή την πρόταση δεν πρέπει μόνο την ασφάλεια της υγείας των ασθενών να προστατεύουμε. Είναι το ανώτατο αγαθό αυτό. Συμφωνώ με την Dagmar Rothberend επ' αυτού. Αλλά δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Θέλουμε να έχουμε λειτουργούσες αγορές. Εκεί όπου θα πολλούνται σε προσιτές τιμές τα φάρμακα να είναι προσιτά σε όλους. Και το καλύτερο φάρμακο δεν ωφελεί αν μόνο σε ένα περιορισμένο κύκλο ασθενών χρησιμοποιείται ή μόνο σε ένα κύκλο ανθρώπων που μπορούν να πληρώσουν απρόσθετες τιμές. Γι' αυτό είναι εξίσου σημαντικό θα έλεγα λειτουργούσες αγορές να δημιουργήσουμε. Και πάλι τα μονοπόλια να κατακαιρματιστούν, να καταπολεμηθούν, ώστε στα κράτη-μέλη στις ε, εταιρείε φαρμακοβιομηχανίες να ανοίξει ο κύκλος των φαρμάκων για όλους. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και ακριβώς στον τομέα της υγείας, ακριβώς αν δει κανείς το δυναμικό αυτών των αγορών, μπορεί να δει ότι πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό υπάρχει, ώστε οι τιμές των φαρμάκων να μειωθούν, να είναι πιο προσιτές. Θέλουμε επίσης με αυτή την πρόταση την ανταγωνιστικότητα την ικανότητα καινοτομία των εταιριών στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία να τις διασφαλίσουμε. Όταν μεγάλα κονδύλια επενδύονται στην ανάπτυξη ενός φαρμάκου, τότε κάποιος θέλει φυσικά να ε, προστατεύει αυτό το φάρμακο με την ευρεσιτεχνία που το καλύπτει. Και εδώ τα προϊόντα μαϊμούδες είναι πολύ βλαπτικά, διότι υπονομεύεται η καινοτομία και αυτό είναι εις βάρος των ασθενών. Αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βέβαια πρέπει να εξετάζεται και όχι μόνο να επικεντρωνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και όλα τα άλλα να τα αγνοούμε. Εδώ θα πρέπει, ας το πω έτσι, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να μην ε, ε, χάσουμε από τα μάτια μας την αντιμετώπιση της ρίζας του κακού. Εδώ ένα σύστημα ασφάλειας να δημιουργήσουμε για τους, ασφαλ... ασθενείς, αλλά ταυτόχρονα και για την φαρμακοβιομηχανία και για τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι σημαντικό, δηλαδή ένα σε ανώνυμο πλαίσιο σύστημα ασφάλειας ε, ε, να μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Όταν δούμε το τι συμβαίνει, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών, Πρέπει να έχουμε υψηλότατες προδιαγραφές ασφάλειας και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θέλω να παρακαλέσω την εισηγήτρια όταν υποβάλει την γραπτή μορφή της έκθεσής της με ένα, ας το πω έτσι να την παροτρύνω, να δείξει μεγαλύτερη γενναιότητα και να ξεπεράσει, ας το πω έτσι, ένα στενότερο πλαίσιο διότι πρέπει να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας και είναι πραγματικότητα αυτή ότι το διαδίκτυο και το εμπόριο στο διαδίκτυο αυτών των φαρμάκων αυξάνεται. Και αν τα δει αυτά και οι απομιμήσεις αυξήθηκαν βέβαια λόγω της ε, πώληση φαρμάκων στο διαδίκτυο. Αλλά χρειάζεται θάρρος, γενναιότητα να το εντάξουμε στις προσπάθειές μας για να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Και έτσι θέλω να ευχαριστήσω και να πω ότι με την προθυμία να συνεργαστούμε μπορούμε να καλύψουμε μεγάλο μέρος της ε, πορείας που πρέπει να ε, καλυφθεί ώστε υπέρ των ασθενών να έχουμε ασφαλή φάρμακα σε προσθέσεις τιμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζήμπερ. Κυρία Λαλής. Είσαστε εδώ. Κυρία Διευθύντρη, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε στα πολύ άριθμα ερωτήματα που ακούσατε. Ελληνίδα είναι αυτή. Ε. Θα ξεκινήσω με τα θέματα της νομικής βάσης, το θέμα των ορισμών, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας το ίντερνετ και δύο λόγια για την επιτροπολογία ολοκληρώνοντας, για την νομική βάση. Η νομική βάση δεν εξαρτάται από τον, τον τόπο της υπηρεσίας κομισιών. Εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης. Μέχρι στιγμής τα φαρμακευτικά ε, καλύπτονταν από το άρθρο 95 και αποφασίζονταν από τους Υπουργούς Υγείας, από αυτή την Επιτροπή, ποτέ από τους Υπουργούς Εσωτερικής Αγοράς ή την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Δεν ε, έχει σχέση δηλαδή αν τα, τα φάρμακα θα περάσουν στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΚΟ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν θα ε, μπορέσουν να εξεταστούν με βάση το άρθρο 168 που είναι το, η νέα ρύθμιση του σημερινού 152. Το άρθρο 168 λέει ότι μπορούμε να αρμονίσουμε την ποιότητα και ασφάλεια των φαρμάκων. Όπως ξέρετε, υπάρχει και μια τρίτη απέτηση για κάθε φάρμακο για να μπει στην αγορά. Και αυτό είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου με βάση το άρθρο 68. Χρειαζόμαστε το 95. Όλα αυτά είναι νομικά θέματα, τα οποία θα ρυθμίσουν οι τρεις νομικές ε, υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων. Το άρθρο 168 ε, έχει και μια δήλωση, τη δήλωση 32 που είναι προσαρτημένη, που θέτει μια νέα προοπτική στο θέμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Υπάρχει μια δοκιμή ε, που θα πρέπει να γίνει για να αποδείξουμε ότι η δημόσια υγεία διατηρείται ε, σε περίπτωση που λαμβάνονται οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό. <clears throat> Αυτή η συζήτηση θα λάβει χώρα αργότερα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε την διτή νομική βάση. Το άρθρο 114, ε, η νέα ρύθμιση του παλιού 95 και το νέο 168. Τώρα για τον ορισμό. Επίσης συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε κάποιους ορισμούς. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του ΠΟΗ. Πάντα υπάρχει όμως μια θεά ζώνη σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Γιατί μπορούμε να έχουμε ένα επιτρεπόμενο νομικό πώς ε, φάρμακο, το οποίο να μην είναι όμως επαρκές. Ε, δηλαδή, ε, κάποιο κουτί, κάποια παρτίδα να, είναι, ε, να μην είναι καλή, χωρίς να είναι α, παραποιημένο. Πάντα θα υπάρχει αυτή η θεά ζώνη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των φαρμάκων. Θεωρούμε όμως ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να ενταχθούν στον ορισμό του κειμένου που συζητάμε σήμερα. Τα θέματα ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση για να καταλάβουμε όλοι το θέμα καλύτερα. Η αυθεντικότητα, η γνησιότητα και η ταυτοποίηση. Αυτά τα θέματα δεν είναι εναρμονισμένα. Αποκλείονται σαφώς από την παρούσα φαρμακευτική νομοθεσία. είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό που θέλουμε την πρότασή μας είναι αυτά τα δύο θέματα να τα εντάξουμε στο εναρμονισμένο πλαίσιο. Προτείνουμε λοιπόν, με βάση τη σημερινή διατύπωση του κειμένου, να έχουμε μόνο ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας και όχι 27 ε, εθνικά συν ένα ευρωπαϊκό. Αυτό λέει το κείμενό μας. Λέει ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας το οποίο θα αντικαταστήσει τα 27 προϋπάρχοντα, αν υπήρχαν. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό λόγω του πεδίου εφαρμογή που προτείνουμε. Προτείνουμε να έχουμε μια προσέγγιση που να βασίζεται στο κίνδυνο. Γιατί θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας στην αρχή της αναλογικότητας. Και όπως εξηγούμε στη μελέτη αντικτύπου, προς το παρόν δεν υπάρχουν ψευδεπίγραφα φάρμακα, ε, παραδείγματος χάρη, ε, που πουλούνται, ε, μιλάω για φάρμακα μη συνταγογραφούμενα. Επομένως, μέχρι στιγμής εστιάζουμε στα συνταγογραφούμενα. Βεβαίως, μπορούμε σε πέντε χρόνια να θεωρήσουμε αυτή την πρόταση. Γιατί μπορεί να αλλάξει το εμπόριο των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις. Τώρα, το χαρακτηριστικό ασφαλείας αυτό δεν κοστίζει. Με βάση τις πληροφορίες μας δεν θα αυξήσει τη τιμή του φαρμάκου. Το θέμα είναι το ζήτημα της ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας και της βάσης δεδομένων. Αλλά ως κοινωνία θα πρέπει να πληρώσουμε το κόστος της ανιχνευσιμότητας των φαρμάκων. Ψάχνουμε τα ίχνη των αυγών, του κρέατος, όχι των φαρμάκων. Είναι κοινωνικό θέμα. Πρέπει να επιλέξουμε ως κοινωνία. Αν δεν θέλουμε να επομιστούμε το κόστος, τότε μειώνεται η ασφάλειά μας. Ε, μειώνεται η ασφάλεια στην αλυσίδα διανομής των φαρμάκων για το ίντερνετ. Κάθε πώληση ενός συνταγογραφούμενου φαρμάκου από, μια, από ένα καναδικό site ε, σε ένα βέλγο κάτοικο, ας πούμε. Παραβιάζει 15 διατάξεις. Υπάρχει ο νόμος. Το θέμα είναι η εφαρμογή του νόμου. Αυτό είναι το πρόβλημα με το ίντερνετ. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες απαγορεύσεις. Υπάρχουν. Απλώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν λόγω της φύσης του ίντερνετ. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να ενδυναμωθεί ο έλεγχος των πωλήσεων μέσω ίντερνετ. Ποιες ιδέες έχετε σύστημα ανείχνευσης, λογότυπου, οτιδήποτε σκεφτείτε, μπορούμε να το σκεφτούμε και εμείς, να το λάβουμε υπόψη μας. Για την επιτροπολογία, ο κύριος Λίσε έθεσε το θέμα. Όταν συντάξαμε αυτή την ε, πρόταση, υπήρχε το θέμα της Πράγας. Τώρα θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Σήμερα? Α, σήμερα κιόλα μπαίνει σε ισχύ. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει η νέα συνθήκη την επιτροπολογία και όλες οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί με βάση αυτή την πρόταση δεξιά και αριστερά, όπως και με τις άλλες προτάσεις. Δεν μπορώ να σας πω τώρα τίποτα πιο συγκεκριμένο για το θέμα της επιτροπολογίας, θα πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ. Το θέμα της επιτροπολογίας με κάνει να σας υπενθυμίσω ότι από τα μεσάνυχτα της 1ης Δεκεμβρίου ήδη ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Να ξαναδώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια. Σίγουρα ακούσατε τα πολλά επενετικά λόγια για την ποιότητα της έκθεσής σας. Οπότε έχετε το λόγο. Ε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θέλω να ευχαριστήσω προφανώς για τις παρεμβάσεις και τα σχόλια και τις προτάσεις που έγιναν και τις αποσαφηνήσεις ε, τώρα στο τέλος που είναι σημαντικό. Πολλή συζήτηση έχουμε μπροστά μας για να συνεχίσουμε. Πολλές συζητήσεις για να προτείνουμε την καλύτερη εφικτή δυνατή λύση ένα πράγμα είναι εκείνο στο οποίο συμφωνούμε σίγουρα όλοι, το σημερινό ε, σύστημα δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα που έχουμε. Και ευχαριστούμε λοιπόν για την ε, ε, υποβολή μιας πρότασης που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας. Ευχαριστώ όλους για το ότι μπόρεσε να είναι εφικτή, δυνατή αυτή η εργασία. Ευχαριστώ. Je vous Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια και όλους εσάς και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την ημερήσια διάταξη πριν κλείσουμε. 25 Ιανουαρίου θα εξεταστεί η έκθεση αυτή. 9 Φεβρουαρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 6 Απριλίου ψηφίζουμε στην Επιτροπή και το Μάιο του 2010 στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και διακόπτη συνεδρίαση. Κύριε Σλούτερ, θέλετε το λόγο. Έχουμε αυτή την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, όπως ξέρετε, και υπάρχει ένα νέο πρόσθετο τροφίμων ε, το οποίο προτείνεται στο παράρτημα του κανονισμού ε961 και θα ήθελα πριν από την λήξη της προθεσμίας, προτάθηκε το Σεπτέμβριο, δηλαδή τέλος Δεκεμβρίου πρέπει να λάβουμε κάποια θέση αν έχουμε αντιρρήσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να το βάλουμε στην ημερήσια λοιπόν, διάταξη, στην ημερήσια διάταξη είτε τώρα είτε για την επόμενη συνεδρία, αλλά να μην χάσουμε την προθεσμία να το συζητήσουμε εγκαίρως. Πρόεδρος. Κύριε Σλούτερ, σας προτείνω να συντάξετε γραπτός μια ένσταση για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε με ανοιχτό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα τα ξαναπούμε στις 3.